ψηφοφορία για αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη θα λάβει χώρα αύριο στι 11 και 30. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του Αντιπροέδρου Πλάσακ όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων των κρατικών ενισχύσεων. Έχετε το λόγο, κύριε Σιγητά. Συνάδελφοι, Πρόεδρε, Επίτροπε, Με το χρόνο που χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προετοιμάσει την πρότασή της, δεν είχαμε και εμείς πάρα πολύ χρόνο να προετοιμάσουμε το δικό μας ε, ψήφισμα, που όμως έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, διότι θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημοκρατικού ελλείμματος ε, στη διαδικασία λήψης ε, αποφάσεων, κυρίως ως προς το πρωτογενές ε, δίκαιο. Συζητήσαμε με τον κύριο Αλμούνια για αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές ως προς την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες αλλαγές που έχουν γίνει ως προς την επιλεξιμότητα των μεγάλων επιχειρήσεων σε παράκτιες σε περιοχές, την τροποποίηση του ποσοστού επιδότησης, τη μειωσή του, δηλαδή επίσης την δυνατότητα χρήσης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, σε παράκτιες περιοχές ε, είναι επιλέξιμες επενδύσεις που γίνονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως διαφωνούμε με την αποτίμηση ε, των επενδύσεων που γίνονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και ενδέχεται να αποθαρρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα είναι πάρα πολύ περίεργο αν διατηρηθούν αυτοί, ε, αυτές οι αλλαγές, ε, διότι ο στόχος ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες ε, των μικρών επιχειρήσεων. Όταν Ε, λοιπόν διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να ορθώσουμε φραγμούς μπροστά στις μεγάλες επιχειρήσεις για να επωφεληθούν οι μικρές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα benchmarking, ένα πίνακα σύγκριση ε, για τη δράση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Παραθέτω τον κύριο Αλμούνια, ε, μας είπε ότι η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική δεν είναι απαραίτητα αλληλοσυμπληρούμενες. Το πρόβλημα είναι ότι Χρησιμοποιούμε διαφορετικά στατιστικά δεδομένα, διαφορετικούς ε, τρόπους χαρτογράφησης και διαφορετικούς ε, κανόνες ε, ανάλογα με το αν εξετάζουμε την πολιτική συνοχή στην περιφερειακή πολιτική και αλλάζουμε τις κλίδες ανάλογα με την πολιτική. Δεν υπάρχει ομοιομορφία δε ως προς την ε, ανάκτηση των κρατικών επιδοτήσεων σε περίπτωση μετεγκατάστασης της επιχείρησης. Ξέρω ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τη συζήτηση για το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, υπολείπονται κάποια σημεία που χρειάζονται εξέταση Δεν έχουμε υπερπηδήσει τις πολιτικές διαφορές, πάντως είναι καθαρά πρακτικά τα προβλήματα και ελπίζω η Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τους σύγχρονη στην κατάσταση. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Σάντζες Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για δεύτερη φορά φέτος επανερχόμαστε σε αυτή τη μεταρρύθμιση για τις κρατικές επιδοτήσεις ε, που αφορούν την περιφερειακή πολιτική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε χωρίς να υπάρχει πραγματική βιωσιμότητα κάποιες ε, επιχειρήσεις Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει εδώ να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Είμαστε κατά της χρησιμοποίησης δημόσιων κονδυλίων για να στηριχθεί η απομάκρυνση επιχειρήσεων από την Ευρώπη. Θεωρούμε πραγματικά ότι αυτές οι δημόσιες επιχορηγήσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Δεν είναι σημαντικό το πόσο μεγάλη είναι μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε μια περιφέρεια, αλλά το πόσο στοχευμένη είναι η δράση της για μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα σε κάποιες διασυνοριακές περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρύβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον ε, κύριο Βλάσεκ. Ήμουν ασκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε πραγματικά υπόψη το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκρίθηκε τελικά θετικά στην εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Ο τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη ανάκαθαν έλεγε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στι πολιτικέ κρατικών ενισχύσεων και, και άλλε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή. Ο κύριος Αλμούνια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ζήτημα αυτό. Θεωρώ πάντως ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω εν ώψη των αλλαγών που γίνονται αυτή τη στιγμή στις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ιδίω στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένου κανόνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κρατικέ ενισχύσει να έχουν απαραίτητους ξεκάθαρου κανόνε και μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου ξεκάθαρου κανόνε. Ευχαριστώ, κύριο Μπάνκι. Excuse me, micro. Το μικρόφωνο σας. Ε, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! A jelentéstevővel egyetértek abban, hogy... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ίσως δεν είναι πολύ κατάλληλη η στιγμή να σταματήσουμε αυτήν την ε, στήριξη κάποιων περιοχών μέσω κρατικών ε, επιδοτήσεων. Εν μέσω κρίσης είναι πολύ σημαντικό το καθήκον των κρατικών αρχών, ο ρόλος των κρατών να στηρίξουν μια δραστηριότητα σε κάποιες περιφέρειες, σε περιφέρειες οι οποίες βεβαίως ε, θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν αυτές τις επιδοτήσεις διότι η οικονομική δραστηριότητα το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού. Το συμφέρον όλων μας είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να ενδυναμωθεί και ενδεχομένως βλέπουμε πότε θα καταργηθούν αυτές οι κρατικές επιδοτήσεις αργότερα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι κρατικέ επιδοτήσει είναι ο πιο άμεσο τρόπο να περικοπεί δημοκρατική συμμετοχή των κρατών μελών. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ω επίθεση κατά τη δημοκρατία για να επιβληθεί η δικτατορία των αγορών. Ε, έχουμε άφθονα κονδυλία τα οποία όμω διοχετεύονται σε μεγάλε πολυεθνικέ επιχειρήσει παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέπει να μετεγκαθίστανται αυτές οι πολυεθνικές λίγα χρόνια μετά τις ε, ε, παχυλές κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν λάβει χωρίς να ανακτά αυτές τις επιδοτήσεις και πλήττονται οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ενώ προσπαθούν να καταπολεμήσουν την απόσταση που τις χωρίζει από τις πιο οικονομικά εύρωστες περιοχές. Χρειάζεται ένα σωστός προγραμματισμός των δημόσιων ε, επιχορηγήσεων και η πράξη έχει αποδείξει ότι ε, δεν συνάδουν αυτοί οι στόχοι ε, με την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι κρατικές επιδοτήσεις όταν χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο μπορούν να επιφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και να τονώσουν την οικονομία της Ευρώπης. Όμως θα πρέπει να κατευθυνθούν προς λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και προς παραγωγικούς τομείς που ενδέχεται να τονώσουν την ανάπτυξη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες με την κρίση. Πρωταρχικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση της ανεργίας των νέων. Αυτά τα εθνικά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο και γι' αυτό υποστηρίζω την απλούστευση των κανόνων σε αυτό το τομέα, καθώς και μια καλύτερη ενημέρωση από πλευράς ε, των δημοσίων αρχών για τις υποχρεώσεις ε, ε, κοινοποίησης, παραδείγματος χάρη σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Εμέτα που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου Βλάσεκ για την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. Η έκθεση αυτή έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη της και τις γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Απασχόλης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να καταφέρουμε δηλαδή να δούμε ποιοι είναι οι κανόνε για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Θέλουμε να προωθήσουμε τι περιφέρειε εκείνε τη Ευρώπη οι οποίε υστερούν και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση βέβαια οι κρατικέ αυτέ ενισχύσει να οδηγήσουν σε στρέβλωση τη εσωτερική αγορά. Θα πρέπει οι ενισχύσει αυτέ να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί κυρίω στι περιφέρειε εκείνε όπου η κρατική ενίσχυση μπορεί πραγματικά να προωθεί στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δώσουν κάποια ποσά χωρί να υπάρχει η εξάντε, ο εξάντε έλεγχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί μια μεγαλύτερη αύξηση των ποσών στις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια στεκτικότητα ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και την πολιτική κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, η αναθόρηση όλων των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες του εξεχρονισμού των κρατικών ισχύσεων θα επιτρέψουν να έχουμε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Η νέα πολιτική όμως συνοχής, καθώς επίσης και η νέα, ο νέος κανονισμός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι δύο διαφορετικές πολιτικές. Θα πρέπει να είναι συνεκτικές αλλά όχι ταυτόσιμες. Ένα άλλο στοιχείο τη μεταρρύθμιση, το οποίο αναφέρεται η έκθεση, είναι η πιο περιοριστική προσέγγιση των ενισχύσεων προ τι μεγάλε επιχειρήσει καθώς επίσης και σε περιοχές της κατηγορίας Γ. Καταλαβαίνετε ότι οι ενισχύσει αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε κακή χρήση των δημοσίων πόρων. Αντίθετα, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2013 και έχοντας ακούσει επίσης και πάρα πολλούς εμπλεκομένους, έχει αποφασιστεί να αυξηθεί ελάχιστα το επίπεδο της γεωγραφικής κάλυψης κατά 45% σε σχέση με αυτό το οποίο προβλεπόταν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προβλέπεται ένα ιδιαίτερο δίκτυο ασφάλειας για τις περιοχές εκείνες που ανήκουν στο πρόγραμμα της μακροπεριφέρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η αύξηση αυτή στην κάλυψη από τις κρατικές ενισχύσεις θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη χρηματοδότησης και κατά αυτόν τον τρόπο δίνουμε το απαραίτητο περιθώριο στα κράτη-μέλη για να καλύψουν ε, περιοχές ε, οι οποίες ε, υστερούν, όπως για παράδειγμα νησιωτικές περιοχές. Η έγκριση των νέων κανόνων προβλέπεται για το δεύτερο ήμιση του Ιουνίου και όπως λέγεται άλλωστε στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει να παρατείνει του υφιστάμενους κανόνες, καθώς επίσης και τη χαρτογράφηση που προβλέπεται αυτή τη στιγμή για τις κρατικές ενισχύσει περιφερειακού χαρακτήρα μέχρι τον Ιούνιο του 2013, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εφαρμόσουν του νέου κανόνες οι οποίοι θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου του 2014 και μετά. Συζητείται πάντως ακόμα το ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένω να γίνει περαιτέρω τροποποίηση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ολοκληρώνουμε με αυτήν την παρέμβαση την συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30 και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο θέμα. Πρόκειται για την έκθεση Higgins, στρατηγική για την υπηρεσία τηλεδιοδίων, σύστημα τελών με